Προχωρούμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Γενοβέφα Γκραμπόφσκα σχετικά με το διάλογο των πολιτών στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας. Τέσσερα λεπτά κυρία Γκραμπόφσκα. Μάικρο, please. I pressed. Thanks. Okay. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επιτροπέ, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε τώρα θέμα και θα μιλήσουμε για τις ε, σχέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών ε, οργάνων ε, και των πολιτών. Εδώ υπάρχουν κενά. Ο Ζαν στο παρελθόν είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΟΚ, τέλο πάντων δεν δημιουργείται για τα κράτη, αλλά για τους πολίτες τους. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχώς διευρύνεται, αλλά τα κοινοτικά όργανα έχουν προβλήματα στην επαφή τους με τους πολίτες. Στο παρελθόν ε, ξέρουμε ότι ε, αυτό οδήγησε σε πολύ ε, θλιπηρά αποτελέσματα το γαλλικό όχι, το ολλανδικό όχι το ιρλανδικό όχι στη συνθήκη της Λισαβόνας οφείλονται ακριβώ αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει η κοινωνία των πολιτών τι, μεγάλη, τι ρόλο παίζει η κοινωνία των πολιτών ε, στον κόσμο μας και στην εποχή μας αλλά ε, τα πράγματα δεν φαίνονται να βελτιώνονται στην επαφή με τα κοινωτικά όργανα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ έχει ένα δικό του ρόλο να παίξει ε, γιατί είναι ακριβώς το όργανο το οποίο θα μπορούσε να ε, βοηθήσει στη μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος. Το άρθρο 10 τις ευρωπαϊκές συνθήκες λέει ότι όλοι οι πολίτες μπορούν να συμμετάσχουν στην λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναλυφθούν πρωτοβουλίες πολιτών με ένα εκατομμύριο υπογραφές οι πολίτες μπορούν να θέσουν ένα ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να πείσουν ενδεχομένως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προετοιμάσει νομοθετική πρόταση. Εγώ στην έκθεσή μου μιλώ για τον διάλογο των πολιτών, ο οποίος βεβαίως δεν ορίζεται στα νομοθετικά κείμενα. Θα ήθελα όμως ο διάλογος αυτός, αν είναι δυνατόν, να ακολουθεί τις εξής αρχές πρώτα πρώτα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό να υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα της κοινωνίας των πολιτών να, να με άλλα λόγια οι συνομιλητές να είναι εκείνοι που πρέπει επίσης ο διάλογος των πολιτών θα πρέπει να είναι αμοιβή να είναι πραγματικός διάλογος όχι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση απλώς να μιλά στον πολίτη και ο πολίτης να καλείται μόνο να απαντήσει να έχει δυνατότητα ο πολίτης να εκφραστεί για να τον ακούσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μας χρειάζεται λοιπόν ένας μηχανισμός ο οποίος ε, τελικά ε, θα εξασφαλίζει αυτό το τον αμφίδρομο αυτόν τον πραγματικό διάλογο Επίσης θα πρέπει ο διάλογος αυτός να ακολουθεί πολύ συγκεκριμένους κανόνες. Δεν ε, θέλουμε να υπάρχει πρόβλημα με το, με ποιος ε, συμμετέχει και όχι ή και ποιος όχι. Βεβαίως όλες αυτές οι αρχές, όλοι αυτοί οι βασικοί κανόνες πολύ δύσκολο να οριστούν. Γι' αυτό περιμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να η οποία τέλος πάντων έχει ασχοληθεί άλλωστε και με το θέμα αυτό ήδη από το 2002 ε, θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, ε, να επεξεργαστεί ενδεχομένως κανόνες, κριτήρια και αρχές που θα πρέπει να γίνονται σεβαστές ε, αυτά που περιλαμβάνονται στην έκθεσή μου Νομίζω ότι είναι θέματα τα οποία θα μπορούσαν κάλλιστα να δοκιμαστούν στις ε, ευρωεκλογές φέτος για να γίνει ένα κάποιο πρώτο βήμα προς τον πολίτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει μια κάποια προσφορά στον πολίτη, να της παρουσιάσει το καλύτερο που έχει. Ευχαριστώ. Η κυρία Βασιλείου. Η Επιτροπή καταρχάς θέλει να ευχαριστήσει την εισηγήτρια κυρία Γκραμπόφσκα και την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων για την εξαιρετική έκθεση. Σύμφωνο ότι η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει έναν καθοριστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ενοποίηση. Είναι ένα από τα βασικά εργαλεία για την επικοινωνία μεταξύ των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κοινωνίας της Ευρώπης και των πολιτών. Βοηθά τους πολίτες να ασκήσουν το δικαίωμά τους να συμμετάσχουν στο δημοκρατικό βίο της Ένωσης. Η Επιτροπή έχει μια μακρά και υγιή παράδοση ε, επικοινωνίας με, τους, ε, με τις οργανώσεις της των πολιτών. Η συνεργασία αυτή μεταξύ Επιτροπής και Κοινωνίας Πολιτών αυξήθηκε και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από τον διάλογο σε θέματα πολιτικής, την διαχείριση έργων, και στο εσωτερικό της Ένωσης και στις χώρες εταίρους. Η συνθήκη της Λισαβόνας θα επισημοποιήσει την υφιστάμενη ε, σχέση μας και θα της δώσει μια περαιτέρω όθεση, ταυτόχρονα δε θα ανοίξει τις πόρτες για την κοινωνία των πολιτών, επιτρέποντας να γίνουν επίσημες οι θέσεις μέσω της λαϊκής πρωτοβουλίας. Ταυτόχρονα Ωστόσο, ο διάλογος αυτός απαιτεί την χορήγηση στην κοινωνία των πολιτών ε, των ενδεδειγμένων εργαλείων για να μπορέσουν να εκφράσουν την άποψη των πολιτών. Γι' αυτό το λόγο ταυτόχρονα και τα όργανα της Ένωσης χρειάζονται τα αντίστοιχα εργαλεία για να είναι σίγουροι ότι αυτά που ακούμε από την κοινωνία των πολιτών και τους πολίτες τοποθετούνται ε, συλλέγονται και τοποθετούν στο σύστημα ως αρμόζει. Η Επιτροπή υποστηρίζει πολλά από τα στοιχεία της έκθεσης, πολλά δε από αυτά τα, έχει ήδη, τα υλοποιεί ήδη. Η Επιτροπή σήμερα έχει αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλειών εμπλοκής των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών σε πολλούς τομείς σε επίπεδα διαβούλευσης για θέματα ένωσης. Ένα από τα πιο καινοτόμα παράδειγμα, παραδείγματα των προσπαθειών αυτών ήταν η διαβούλευση με τους πολίτες και η ε, διεπικοινωνιακή ε, συζήτηση. Για να καταλάβουμε τις ανάγκες των πολιτών, αναπτύξαμε τα τελευταία 35 χρόνια το Ευρωβαρόμετρο, που αποτελεί πλέον ένα εξαιρετικά ε, πολύτιμο εργαλείο για την παρακολούθηση της κοινή γνώμης στην Ευρώπη. Αλλά ούτε η Επιτροπή, ούτε το Κοινοβούλιο μπορούν μόνοι τους να δημιουργήσουν και να οργανώσουν μια, ένα πανευρωπαϊκό διάλογο. Τούτο θα καταστεί δυνατό μόνο όταν συνεργαστούν τα εθνικά, τα κράτη-μέλη και τα ευρωπαϊκά όργανα και αυτός ήταν ο στόχος της ε, ανακοίνωσης και της διοργανικής συμφωνίας που είχαν υπογράψει στις 22 Οκτωβρίου του 2008 τα τρία μεγάλα θεσμικά όργανα και με τον τίτλο επικοινωνώντας με τους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο συντονίζουν ήδη τι προσπάθειε του με τα κράτη-μέλη μέσω τη διαχείριση εταιρικών σχέσεων που περιλαμβάνουν τοπικέ και περιφερειακέ καμπάνιες για συγκεκριμένα θέματα που ε, παρακολουθούν και συνδέονται με αντίστοιχε δράσει, ΜΚΟ και τοπικών πρωτοβουλειών. 11 νέε εταιρικέ σχέσει αυτή τη μορφή το 2009 θα καταστήσουν ακόμα αποτελεσματικότερη την προσέγγιση αυτή. Συμφωνούμε ως Επιτροπή με την άποψη ότι ο καρποφόρος διάλογος εξαρτάται από την ενεργό συμμετοχή όλων των πλευρών, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, των κρατών μελών και της κοινωνίας των πολιτών. Η Επιτροπή ελπίζει ότι η συνθήκη της Λισαβόνας θα τεθεί σε ισχύ και είναι έτοιμη να αναλάβει την αναγκαία δράση για να υλοποιήσει τις διατάξεις της και να συνεχίσει να αναπτύσσει τον διάλογο με τους πολίτες. Ευχαριστώ. Thank you. Eh, eh? Αύριο θα ψηφίσουμε. Η έκθεση που είχαμε προβλέψει να συζητηθεί από την κυρία Ντοϊκένε δεν θα συζητηθεί γιατί λείπει. Θεωρούμε ότι παρουσιάστηκε ωστόσο και θα ψηφιστεί την Τετάρτη. Είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό η ανάπτυξη του Συμβουλίου των